και την προσωπική μου και εν ονόματι του Πρόεδρου Σούλτς. Θέλω να σας πω ότι η γραπτή δήλωση των συναδέλφων Αλμπερτίνη, Νικολάς Μπερβίσκα, Ρινάλντι και Σασόλη σχετικά με τη στήριξη για μια Ευρωπαϊκή ημέρα για την ε, μνήμη των δικαίων έχει την στήριξη της ε, πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου και θα μεταδοθεί και θα δημοσιευθεί στα πρακτικά αυτή της ε, συνεδριάσεως. Ο κύριος Αλμπερτίν είναι ο πρώτος που υπέγραψε αυτό το κείμενο. Κύριε Πρόεδρε, ε, θέλω να θεωρήσω ότι ε, έπρεπε ε, να υπάρξει ένα μια, ένα κληροδότημα της ανθρωπότητος στους Εβραίους οι οποίοι ε, είχαν ε, σκοτωθεί και ε, πρέπει να υπάρξει και μια ανάμνηση για το μακελιό της Αρμενίας υπάρχουν και άλλες τέτοιες περιπτώσεις δεν πρέπει να τις απλοποιούμε και χρειαζόμαστε ένα πραγματικό παράδειγμα σχετικά με την συμμετοχή ή όχι σε ε, γενοκτονίες. Οι ε, άνθρωποι οι οποίοι με δικό τους προσωπικό κίνδυνο έχουν αντιταχθεί σε τα περιστατικά αυτά συμβάλλουν στην ηθική ανάταση του αισθήματο των ευρωπαϊκών λαών. Ζητώ λοιπόν να ψηφίσουμε τώρα. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Έχετε ψηφίσει όλοι.